Έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Από την ομάδα του ΕΛΚΑ μου έχει ζητηθεί να ορίσουμε την Ελίζα Μωρίν Τσάρτιερ ως μέλος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Δύο Φύλων. Σχόλια από αυτού. Ο ορισμός λοιπόν εγκρίνεται.